Το 2015 θα έχουμε τη νέα περίοδο της κοινή γεωργικής πολιτικής. Επομένως, το 2014 είναι ένα έτος μεταβατικό. Από χρηματοοικονομικής όμως πλευράς ελπίζω ότι μέχρι τον Ιούλιο θα μπορέσει να αρχίσει να ισχύει η συμφωνία αυτή την οποία θέλουμε, στην οποία θέλουμε να καταλήξουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο. Ο Σέρτζο Σιλβέστρης έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρο. Κοιτάξτε, ο George Λάιον με κάλυψε κατά κάποιο τρόπο. Συμφωνώ απόλυτα με τα όσα είπε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την Αν Γένσεν για την παρουσίαση την οποία μας έκανε. Ωστόσο, το ερώτημα το οποίο μας απασχολεί αυτή τη στιγμή, το ζήτημα το οποίο μας απασχολεί δεν είναι εύκολο. Το 2014 θα έχουμε μια κοινή γεωργική πολιτική η οποία ουσιαστικά θα αποτελεί μια επέκταση των όσων ισχύουν για το 2013 με μία μείωση μάλιστα των πόρων. Αυτό θεωρώ ότι δεν είναι ιδιαίτερα λογικό. Επίσης, το να θεωρούμε ότι ε, η γεωργία αποτελεί ένα είδος ε, τραπεζικού ATM, όπου κάθε φορά πηγαίνουμε και παίρνουμε χρήματα από εκεί, αφαιρούμε χρήματα τελικά από τον προπολογισμό για τη γεωργία για να κάνουμε άλλα πράγματα, είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να δεχτούμε. Μου φαίνεται παράλογο ότι ακόμα και στη συζήτηση που είχαμε στην Ολομέλεια, ο Επίτροπος Τσόλος ο ίδιος θεώρησε δεδομένο το ότι ε, οι κοινοτικοί πόροι για τη γεωργία θα πρέπει να περικοπούν ο Τσόλος ε, τελικά με ποια πλευρά ουσιαστικά βρίσκεται ή συμμετέχει τελικά στην ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως Επίτροπος Αρμόδιος για γεωργικά θέματα, γνωρίζοντας ότι απλώς υπάρχουν εκεί κάποιοι διαθέσιμοι πόροι που μπορούν να περικοπούν. Επίσης, κάθε φορά που τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα έχουν μια νέα υπηρεσία, η οποία απαιτεί βέβαια και μια νέα χρηματοδότηση, ουσιαστικά χρησιμοποιούν πόρους από τη Γεωργία για να χρηματοδοτήσουν την νέα αυτή υπηρεσία. Έχουμε για παράδειγμα το, την ύπατη εκπρόσωπο για την εξωτερική πολιτική και χρησιμοποιήθηκε χρηματοδότηση για τις αρμοδιότητες της ύπατου εκπροσώπου για το γραφείο της και καθεξής από την Γεωργία. Πάντως θα πρέπει να συντοποιούμε ότι οι γεωργικές υπηρεσίες είναι εξίσου σημαντικές. Είτε πρόκειται για τη γεωργία του παρελθόντος, είτε πρόκειται για τη σημερινή γεωργία. Αυτό το οποίο βλέπουμε όμως είναι ότι μειώνονται όλο και περισσότερο οι πόροι της γεωργίας και καλούμεθα όμω να επιτελέσουμε ακριβώ τι εργασίε στα πλαίσια τη γεωργία. Οι στόχοι μα και οι προσδοκίε μα παραμένουν οι ίδιε και παρόλα αυτά μειώνουμε συνεχώ την χρηματοδότηση που δίδεται στη γεωργία. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε του πόρου τη γεωργία για να χρηματοδοτούμε άλλε υπηρεσίε και άλλε δραστηριότητε. Επίσης, συμφωνώ με τα όσα είπε ο George Lyon. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να δούμε πώς θα διαχειριστούμε τη μεταβατική αυτή φάση χωρίς χρήματα. Το 2014 θα είναι ένα έτος κατά το οποίο θα πρέπει να αρχίσει να, μάλλον θα πρέπει να συνεχιστεί η, ο κανονισμός αυτός για την κοινή γεωργική πολιτική, ο οποίος ξεκίνησε το 2013. Πώς θα καταφέρουμε να το πράξουμε όμως αυτό όταν θα έχουμε περικομμένους πόρους. Φοβάμαι ότι δεν θα καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε μια βεβαιότητα τόσο για τους ίδιους τους γεωργούς όσο και για εμάς στο ευρωπαϊκό επίπεδο, ότι θα καταφέρουμε δηλαδή να επιτελέσουμε και να συνεχίσουμε τη γεωργική πολιτική. Πρόεδρος. Ευχαριστούμε Σέρτζιο. Αν δεν υπάρχουν άλλοι ομιλητές, να ξαναδώσω το λόγο στην Αν Γένσεν και στη συνέχεια θα ακούσουμε τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα ολοκληρώσει από τη ζήτηση αυτή η Ντάνσιλα. Ε, yes, Ευχαριστώ πολύ. Κάποιες από τις ερωτήσεις πρέπει να κληθεί η Επιτροπή να τις απαντήσει, πιστεύω. Αλλά πάντως, εάν μιλάμε για σίγουρα πράγματα και πράγματα που δεν είναι σίγουρα. Εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία και παραμείνουμε στο σύστημα του 2013, τότε οι μεμονωμένε πληρωμέ θα είναι αυτέ οι οποίε θα μείνουν ενισχύει, τα πόνα κονδύλια δηλαδή τα οποία θα καταβάλλονται στου γεωργού. Αυτή είναι η μόνη βεβαιότητα. Είδαμε όμω και με τη δημοσιονομική πειθαρχία και με τα νέα όρια, ανώτατα όρια ότι υπάρχουν στοιχεία αβεβαιότητας. Ο κύριος Σιλβέστρης ανέφερε ότι η κοινή γεωργική πολιτική είναι σαν ένα τραπεζικό ATM του προϋπολογισμού σε αυτή την προγραμματική περίοδο και έχει δίκιο, διότι όταν ε, προβλέφθηκε το πολιτές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο 2007-2013, μέσα στη νύχτα φρόντισαν να θέσουν πολύ, πολύ ψηλά ποσά στην αρχή της προγραμματικής περίοδου, σταδιακά μειώνοντας τα, ενώ ήταν γνωστό και το έχουμε συστήσει και στην Επιτροπή σας εδώ, ότι θα μειώνονται τα ποσά με το πλησίασμα και τη δημοσιονομικής πειθαρχίας, γιατί είναι όλο και πιο μικρό το περιθώριο. Και αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο ε, χρησιμοποιούμε από την γεωργική πολιτική τα περιθώρια που έχουμε για άλλα προγράμματα, το Γαλιλαίο, τις εξωτερικές σχέσεις. Αυτό όμως δεν θα ξανασυμβεί στη νέα προγραμματική περίοδο. Φτάνουμε πιστεύω σε ένα στάδιο και Φαίνει καθήκον της Επιτροπής σας πιστεύω, ε, φτάνουμε σε ένα επίπεδο που πια τα ποσά που αφιερώνονται στη γεωργία είναι πολύ περιορισμένα, με πολύ περιορισμένο περιθώριο και πρέπει να καταστεί φες ότι δεν μπορεί κανείς να αντλεί ποσά από τον προπολογισμό της γεωργίας. Γι' αυτό χρειάζεται μια γενικότερη ευελιξία. Η ευελιξία όμως θα πρέπει και να συνεπάγεται πως κονδύλια που δεν έχουν απορροφηθεί θα μπορούν να δαπανηθούν σε άλλους τομείς. Και θα βρεθείτε σιγά σιγά σε μια κατάσταση όπου η δημοσιονομική πειθαρχία θα διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο. Αυτό το πώς δηλαδή θα του χειρίσει το θέμα αυτό πρέπει να το απαντήσει και να το εξηγήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά πιστεύω ότι και η Επιτροπή σας θα πρέπει να τοποθετηθεί ξεκάθαρα. Συμφωνώ με αυτά που άκουσα από την εισηγητριά σας και για το ζήτημα των επαρκών ποσών. Ιδιαίτερα θέμα που αφορά την Περιφερειακή Επιτροπή αλλά και στην ανάπτυξη της υπαίθρου έχει πολύ μεγάλη σημασία να έχουμε αρκετά κονδύλια στη θέση μας για να ε, υπηρετούμε, να ε, εξυπηρετούμε καλύτερα τις πληρωμές. Ευχαριστώ πολύ για τα σχόλια. Τα παίρνω μαζί μου, τα μεταφέρω και βέβαια περιμένω να ακούσω η Επιτροπή πώς θα απαντήσει στο θέμα των πληρωμών. Ευχαριστούμε. Έστρε Ντελάντζ έχει ζητήσει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σα ζητώ συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη και από την εισηγήτρια για την καθυστέρηση αυτή, μολονότι είμαι χριστιανοδημοκράτης, δεν καταφέρνω να βρίσκομαι σε δύο μέρη την ίδια στιγμή. Χρειάστηκε λοιπόν να τρέξω γρήγορα από μια άλλη συνεδρίαση. Η βοηθό μου με ενημέρωσε συντόμω για τα ζητήματα τα οποία συζητάτε. Θα ήθελα να προσθέσω δυνατόν δύο συγκεκριμένα ζητήματα. Προφανώ ε, η εισηγήτρια αναφέρθηκε στα πιλωτικά προγράμματα και τι προπαρασκευαστικές δράσει. Θεωρώ παραδοσιακά αυτό που είναι σημαντικό την Επιτροπή μας είναι να ασκούμε πίεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τα περιθώρια τα οποία μπορούμε να έχουμε, τα χρηματικά. Ιδίως όσον αφορά το παρατηρητήριο, όλο και περισσότερες πληροφορίες χρειαζόμαστε από το εφιστάμενο πλέον αυτό σύστημα, το οποίο όμως επικεντρώνεται ιδιαίτερα στις ε, τιμές των ε, αγροτικών προϊόντων στο αγρόκτημα και στο σούπερ μάρκετ, αλλά δεν γνωρίζουμε τελικά τι γίνεται με τις τιμές στα ενδιάμεσα στάδια της αλυσίδας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θυμηθείτε τι λέγαμε χθε με τον Επίτροπο Μπαρνιέ. Λέγαμε ότι υπάρχουν διάφορες αθέμητες πρακτικές, οι οποίες ε, εμπλέκονται τελικά σε όλους τους διαμεσολαβητές ανάμεσα στην παραγωγή και την τελική κατανάλωση, σε όλη δηλαδή την τροφική αλυσίδα. Είναι πολύ σημαντικό να ασχοληθούμε λοιπόν και με το ζήτημα αυτό. Δεύτερο ζήτημα. Εγώ θα καταθέσω, όπως το έκανα και στο παρελθόν, μία τροπολογία προκειμένου να αυξηθεί λίγο ο προπολογισμό για την υπηρεσία, την, ιατρική και την αρμόδια για τα τρόφιμα. Πρόσφατα είχαμε το σκάνδαλο με το κρέας αλόγου, το οποίο παρουσιαζόταν ως βόλιο κρέας βλέπουμε όλο και περισσότερες παρατυπίες ή απάτες στο πλαίσιο των τροφίμων. Μάλιστα η Επιτροπή Περιβάλλοντος θα καταθέσει μία έκθεση πρωτοβουλίας για το ζήτημα αυτό, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει όλο και περισσότερο έντονο το φαινόμενο αυτό της τροφικής απάτης το πρόβλημα είναι ότι βλέπουμε όλο και περισσότερε νέε περιπτώσει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να δούμε πώ μπορούμε να αυξήσουμε κάπω τον προπολογισμό τη κτηνιατρική τροφική υπηρεσία, προκειμένου οι υπάλληλοι του γραφείου αυτού να φύγουν από τα γραφεία του και να καταφέρουν να κάνουν όλο και περισσότερου επιτόπου διερευνητικού ελέγχου και μάλιστα χωρί να του ανακοινώνουν εκ των προτέρων. Νομίζω ότι κάνοντας κάποια εξοικονόμηση στις άλλες υπηρεσίες θα καταφέρουμε να πρημοδοτήσουμε περισσότερο αυτή την υπηρεσία. Δεν θεωρώ ότι είναι δεδομένο αυτό, αλλά καθότι βλέπουμε όλο και περισσότερες περιπτώσεις τροφικής απάτης, θεωρώ θα πρέπει να ασχοληθούμε και αυτό. Και πλήττεται κυρίως ο πρωτογενής τομέας, ο οποίος δεν ευθύνεται βέβαια για την απάτη αυτή, η οποία γίνεται κάποια στιγμή αργότερα στη διατροφική αλυσίδα και όχι στο αρχικό στάδιο. Δύο συγκεκριμένα λοιπόν ζητήματα που θέλω να θέσω αυτά και μία παρατήρηση. Ελπίζω ότι αυτή τη φορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιτέλου θα θέλει τα χρήματα. Γιατί όταν έκανα ανάλογη πρόταση πριν από μερικά χρόνια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μα είπε όχι, όχι, όχι πολύ ε, θετικό το ότι προτείνεται μία αύξηση για την υπηρεσία αυτή, αγαπητό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν τη θέλουμε. Όταν μου λέτε όμως τέτοια πράγματα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ουσιαστικά είναι σαν να μου λέτε ότι δεν σας ενδιαφέρει να εντείνετε τους ελέγχους. Είναι σαν να μου λέτε ότι ας είναι Ευρωπαϊκή νομοθεσία, αλλά ας κάνουν τον έλεγχο μόνο τα κράτη-μέλη, ότι είναι αποκλειστικά εθνική τους αρμοδιότητα. Αν πραγματικά πρεσβεύεται κάτι τέτοιο, θεωρώ ότι πραγματικά υπονομεύουμε τη δική μας την ευρωπαϊκή αρμοδιότητα εδώ πέρα. Δεν μπορούμε να εγκρίνουμε ευρωπαϊκέ νομοθεσίε και στη συνέχεια να μην ασχολούμεθα με τον έλεγχο τη εφαρμογή νομοθεσία αυτή σε εθνικό επίπεδο. Ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δείξει μια πιο επεύθυνη στάση αυτή τη στιγμή και πραγματικά να ζητήσει και αυτή αύξηση των προπολογισμών για να γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι. Ευχαριστούμε πολύ, Έστερ. Αν δεν υπάρχουν άλλοι ομιλητέ, σα ακούσουμε τον εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την DG Agri, Κριστίνα Μόρτσι, διευθύντρια. Είναι εδώ παρούσα και θα ολοκληρώσει η Ντάνσιλα στη συνέχεια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να κάνω δύο σχόλια την δημοσιονομική πειθαρχία. Σωστά, η δήλωση της Επιτροπής για την ε, προτάσεις μεταρρύθμισης κάπου βασίζεται στις προτάσεις του πολιετούς ήδη απέδειξε ότι για το 2014 οι εκτιμήσεις τότε ήταν ότι θα υπάρξει δημοσιονομική πειθαρχία που πρέπει να εφαρμόσουμε. Επίσης, επιτρέψτε μου να σας πω ότι ο κανονισμός τη μεταβατική περίοδο την οποία εσείς και το Συμβούλιο πέρσι συμφωνήσατε για τις άμεσες πληρωμές αφορούσε το 2013 και είπαμε ότι θα εφαρμοστεί και για το 2014. Άρα για τον προπολογισμό που τώρα αρχίζουμε να συζητούμε για του χρόνου. Τώρα, όσον αφορά τη δημοσιονομική πειθαρχία, η Επιτροπή από την επόμενη εβδομάδα, από την 21η Μαρτίου, πρέπει να σας προτείνει και στο Συμβούλιο και σε εσά πώς θα εφαρμοστεί στα πλαίσια του προπολίου του 2014, δημοσιονομική πειθαρχία. Ετοιμάζουμε την, επιτροπή μας, την ε, πρότασή θα φτάσει σε εσά την επόμενη εβδομάδα, διότι η προθεσμία είναι 31η Μαρτίου και μετά και εσείς και το Συμβούλιο θα πρέπει να αποφασίσετε ποσοστά μέχρι τέλος του Ιουνίου. Εάν λοιπόν μέχρι τις 30 Ιουνίου δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ ημών και του Συμβουλίου θα αποφασίσει για το ποσοστό η Κομισιό και αργότερα μες στο έτος θα προτείνει προσαρμογή και στα πλαίσια της ε, τροποποιητικής ε, επιστολής όταν θα ξέρουμε πώς έχουν διαμορφωθεί οι δαπάνες της ΚΑΠ και τότε στα πλαίσια του πολιετούς θα προτείνουμε το σωστό ποσοστό και μπορείτε εσείς μόνο ως Κοινοβούλιο μέχρι την 1η Δεκεμβρίου επίσης να κάνετε αναπροσαρμογή. Γιατί 1η Δεκεμβρίου, διότι όπως είπε σωστά η συγγήτρια, στην 1η Δεκεμβρίου θα αρχίσουμε να καταβάλουμε τα ποσά για τις άμενες πληρωμές. Και τα κράτη-μέλη και οι αγρότες θα πρέπει να ξέρουν τότε ποιο είναι το ποσοστό. Αυτά μπορώ να σας πω για τη δημοσιονομική επιθαρχία. Θα υπάρξει πρόταση και βεβαίω θα τη λάβετε εσείς και εσείς θα πρέπει να τη συζητήσετε. Ευχαριστώ. Αν δεν θέλει κανείς άλλο το λόγο. Η Βιορίκα. Άκουσα με προσοχή τι είπαν οι συνάδελφοι και κυρίως είδαμε ότι θα πρέπει να υπάρχει το γιατί κάνουμε. Όλοι όμως είπανε ότι θα πρέπει οτιδήποτε κάνουμε να ε, έχει ως στόχο ότι οποιαδήποτε πρόταση αφορά μείωση θα πρέπει να την απορρίψουμε. Ξέρουμε ότι τους στόχους τους θα τους υπερασπιστεί η Κομισιό και εμείς θα πρέπει να δούμε πώς θα κάνουμε τη διασύνδεση μεταξύ του δικού μας προπολογισμού, της μας, του κονδυλίου που αφορά τη δική μας την Επιτροπή και αυτή που αφορά γενικότερα τον προπολογισμό όλου του Κοινοβουλίου του 2014. Απλώς μία διευκρίνηση συμπληρωματική από την Κομισιό. Μας είπατε ότι θα έχουμε φέτος την δημοσιονομική πειθαρχία. Τι σημαίνει αυτό ότι θα υπάρχει μία μείωση 2-3% όσον αφορά τις άμεσες ε, πληρωμές μεταξύ των κρατών μελών. Πώς ακριβώς, πώς ακριβώς αυτό το 2-3% ε, θα λειτουργήσει, μπορείτε να μας το εξηγήσετε. Ευχαριστώ. Η Κομισιόν και πάλι ζητάει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτό το οποίο θα κάνει η Επιτροπή σύμφωνα με τον κανονισμό της άμεσης πληρωμές είναι να καθορίσει ένα ποσοστό που θα πρέπει να εφαρμοστεί για τους αγρότες. Όχι για τα κρατημέλη, για τους αγρότες, τους οποίους, ποσοστό το οποίο θα πρέπει να εφαρμόσει κάθε κράτος μέλος κάνοντας τον υπολογισμό για κάθε αγροτική εκμετάλλευση, για κάθε αγρότη. Όπως σας είπα, μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας θα σας ανακοινώσουμε αυτό το ποσοστό. Ευχαριστώ η κυρία Μαγκίνες. Μία περαιτέρω διευκρίνηση. Αυτό το ποσοστό θα ισχύει για όλους τους αγρότες, όποιο και να είναι η ε, αγροτική τους εκμετάλλευση ή το μέγεθος έχει κάποια διαφορά. Η Κομισιά. Και πάλι, οι προτάσεις της Επιτροπής θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Απλώς θα ήθελα να πω ότι το 2003 όταν υιοθετήθηκε η μεταρρύθμιση είχε πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι το όριο του 5.000, στο 5.000 ευρώ θα ίσχυε και για την δημοσιονομική πειθαρχία και για την πολλαπλή συμμόρφωση. Και οι προτάσεις του άρθρου 8 για την επόμενη περίοδο πάλι προβλέπουν 5.000 ευρώ ω όριο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά πάλι αυτά, όπω είπα, την επόμενη εβδομάδα θα υιοθετηθούν οι προτάσει από Επιτροπή. Μάλιστα. Αγαπητοί συνάδελφοι, αν δεν υπάρχουν άλλοι που θέλουν να πάρουν το λόγο, μπορούμε να ολοκληρώσουμε στο σημείο αυτό τη συνεδρία τη Επιτροπή μα. Σα υπενθυμίζω ότι ε, θα συνεδριάσουμε πάλι στι 25 Μαρτίου στι 3 το μεσημέρι. Και θα ήθελα να ζητήσω από του συντονιστέ να παραμείνουν στην αίθουσα για να ολοκληρώσουμε το τμήμα εκείνο τη συνεδρίασής μα που δεν καταφέραμε να, καλύψουμε σήμερα το πρωί. Λύεται συνεδρίαση.